Χαίρετε. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια σύντομη ψηφοφορία σήμερα. Ας αν έχετε τις κάρτες σας να κάνουμε μια επαλήθευση, μια δοκιμαστική ψηφοφορία, όποιο κουμπί θέλετε πατήστε, μόνο και μόνο για να δούμε ότι είστε εδώ. Κυρία Μπορζάν, ψηφίζετε εσείς. Ωραία, πολύ καλά και σας ευχαριστώ. Αρχίζουμε την ψηφοφορία, δημοσιονομικός έλεγχος, ε, χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Με συγκίτρια την κυρία Τόρνανό, τροπολογία 6, ξεκινούμε υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 8 υπέρ κατά απόχέ, απεριφθεί υπέρ κατά απόχέ απεριφθεί 12 ε, 11 συγγνώμη α όχι είχε συρθεί. 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 16 δύο τμήματα Πρώτο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 15 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 15. Άρχεται. Πέρας. Καλώς. Ε, πείτε μας πώς θέλετε να ψηφίσετε. Κατά. Ωραία. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας λοιπόν και εγκρίνεται. Πού ήμασταν 17 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά επαληθεύουμε αρχής ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απερίφθη δεύτερο υπέρ όχι έχει καταπέσει με την απόρριψη μάλιστα και άρα πάμε στην 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30-31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Η 33 έχει αποσυρθεί. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Η 35 έχει αποσυρθεί. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 44 υπέρ απερίφθη, έχει αποσυρθεί μάλλον 45 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 47 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 48 σε πρώτο σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Προλάβατε. Ωραία. Εγκρίνεται. Σαράντα εννέα λοιπόν τώρα. 41 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 50 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 54 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 57 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 60 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 61 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 62 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 63 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 64 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ Κατά. Καταπίπτει. Όχι. Το ψηφίζουμε το δεύτερο. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Δεύτερη υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τρίτη υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τέταρτη απεσύρθη. Πέμπτη υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη και τελική ψηφοφορία ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Okay, Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη συζήτηση σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πρώτο θέμα σήμερα την εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για μακρύτερη διάρκεια ζωής προϊόντων με την κυρία Μόζερ. Και σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Ah, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, κοιτάξτε, λίγο όμως να ησυχάσει η αίθουσα έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ ε, να ε, μιλήσω. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά στην ε, Επιτροπή μας εγώ παρουσίασα το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο αφορά την διασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των προϊόντων. Πρέπει να σας πω ότι το προσχέδιο της έκθεσής μου βασίζεται κυρίως ε, σε μια σειρά παρατηρήσεων ε, που αφορούν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα επικινθεί ε, η ζωή αυτών των προϊόντων. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να το συζητήσουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πιο βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την πραγματικά κυκλική οικοδομία, πώς να έχουν τα προϊόντα μας ε, μακρότερο βίο ε, και επίσης ε, πώς να βοηθήσουμε το περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Εγώ παρουσιάζω αυτό το θέμα με μεγάλη ευχαρίστηση γιατί είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα κατάλογο των προτάσεων είτε προέρχονται από τις επιχειρήσεις, από τους καταναλωτές, από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι αυτές οι προτάσεις για την εξασφάλιση μακρύτερης ζωής ε, των προϊόντων μας. Κυρίως, κυρίως η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει μεγάλη, ε, μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δηλαδή η περιβαλλοντική διάσταση του θέματος πολύ μεγάλη. Είναι σημαντικό λοιπόν να κινητροδοτήσουμε ε, αυτήν την ε, προσπάθεια. Ε, όταν αναφερόμαστε σε οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να δώσουμε και νέα υποδείγματα για αυτήν την οικονομική ανάπτυξη. Δεν μιλάμε μόνο για καινούρια προϊόντα. Θέλουμε εδώ να αναφερθούμε για προϊόντα τα οποία θα παράγονται με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, η Σουηδία μόλις ε, ε, μείωσε τον ΦΠΑ για την επισκευή προϊόντων. Μπορεί να είναι ακόμα και παιχνίδια. Μιλάμε για διαφόρων ειδών προϊόντα. Ε, ε, δηλαδή με τον τρόπο αυτό να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα προϊόντα αυτά. Είναι σημαντική η χρήση και η επανάχρηση των προϊόντων και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εμπνευστούμε από τις χώρες αυτές οποίες έχουν προχωρήσει περισσότερο και οι οποίες δίνουν κίνητρα για την ε, επισκευή ε, προϊόντων καθημερινής χρήσης. Ε, απ' την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι αυτή η σουηδική πρωτοβουλία δημιουργεί και θέσεις εργασίας, ακριβώς λόγω του ότι δημιουργούνται πλέον φορείς που επισκευάζουν τα παιχνίδια. Θα πρέπει να εγγυηθούμε μεγαλύτερη ζωή των προϊόντων και δεν θα πρέπει να το δούμε μονάχα μονάχα από φορολογική και νομική πλευρά. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το design τους, δηλαδή τη στιγμή που τα προϊόντα, τα νέα προϊόντα σχεδιάζονται, θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επισκευαστούν. Επομένως, ε, η Κομισιόν ε, θα πρέπει να επιβάλλει και κάποιες ε, υποχρεώσεις. Ας πούμε, μέσω της οδηγίας για τις μπαταρίες θα πρέπει να, ηλεκτρικές στήλες δηλαδή και συσσωρευτές, θα πρέπει να δίνεται ή να αναλαμβάνει ο κατασκευαστής κατασκευαστή στην υποχρέωση να σχεδιάζει τα προϊόντα με τρόπο έτσι ώστε να καθιστά δυνατή την αντικατάσταση των ε, ηλεκτρικών στυλών. Επίση, ε, μπορεί κανεί να σκεφτεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν και κάποιε περιβαλλοντικέ ε, υποχρεώσει. Πρέπει να συμφωνούμε όλοι γιατί κάποια προϊόντα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πλέον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στη φύση. Επομένως με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ε, και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στις ε, δηλώσεις μας, ε, έτσι ώστε να κινητροδοτήσουμε και τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν περισσότερο τα προϊόντα τους, ενδεχομένως μέσω μιας ετικέτας που θα δίνουν, ε, μια ετικέτα που θα δίνει πληροφορίες και για τη διάρκεια ζωής ας πούμε για το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι σημαντικό ο καταναλωτής να έχει σαφή και συγκεκριμένη ιδέα ε, για την ε, διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, να ξέρει τι τον περιμένει. Αυτό είναι ε, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να παίζει ρόλο στην απόφαση που θα πάρει ο καταναλωτής αν θα αγοράσει ή όχι το προϊόν. Τη στιγμή της αγοράς δηλαδή θα πρέπει να ξέρει ότι έχει και αυτή την δυνατότητα να προστατέψει το περιβάλλον. Βεβαίως βεβαίως ε, πολλά συγκεκριμένα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, πολλά πρακτικά στοιχεία μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην ε, εργασία μας έτσι ώστε ας πούμε αυτός ο κατάλογος των ιδεών που ανέφερα προηγουμένως να διασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ε, σε μια σειρά προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό και θα αποταμιεύσουμε ε, οικονομικά, δηλαδή και η τσέπη μας ε, θα ωφεληθεί αλλά κυρίως θα ωφεληθεί το περιβάλλον και θα έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης, ένα είδος ανάπτυξης το οποίο δεν θα βασίζεται στη διαρκή και ανανέωση των προϊόντων και στην ε, ε, άκρατη και άκρητη κατανάλωση. Υπενθυμίζω ότι εμείς εδώ ως Επιτροπή Περιβάλλοντος οφείλουμε πάντα να βλέπουμε, να συνυπολογίζουμε την περιβαλλοντική διάσταση ε, στις ε, εκθέσεις μας. Ε, και επομένως να σας πω ότι μέχρι τις 18 Μαρτίου μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Έχετε χρόνο έτσι ώστε να υποβάλλετε τροπολογίες γιατί στις 11 Απριλίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μετά στις 24 Απριλίου θα έχουμε την τελική ψηφοφορία. Ευελπιστώ σε ε, στην καλύτερη δυνατή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ωραία. Τώρα θα γίνει ο γύρος των σκιωδών. Η κυρία Κόλιν Λάγκεν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστώ καταρχάς την Κριστέα Σχαλδεμούτσερ για την εκθεσή της, η οποία αποτελεί, πιστεύω, μια πολύ καλή βάση συζήτησης και χαίρομαι ιδιαίτερως για ε, την ευκαιρία αυτή για συνεργασία. Τα οικολογικά πλεονεκτήματα της έννοιας ε, της ε, μεγαλύτερης διάρκειας ζωής για τα προϊόντα είναι αυτονόητα, διαρκούν περισσότερο τα προϊόντα, δεν χρειάζεται να τα αντικαταστήσουμε τόσο γρήγορα, δεν παράγουμε περισσότερα σκουπίδι και εξοικονομούμε και την ενέργεια την απαραίτητη για την παραγωγή των προϊόντων. Θα συμφωνήσω λοιπόν με την εισηγήτρια ότι ιδιαίτερα πρέπει να μιλήσουμε για την βιώσιμη παραγωγή και τα πλεονεκτήματα μιας ε, κυκλικής οικονομίας πρέπει να προέρθουν από την εξοικονόμηση και στην παραγωγή, το κόστος παραγωγής, την άρια παραγωγής και τελικά την κατανάλωση. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερως για το ότι έχει και την παράταση ζωής αλλά και την αποτελεσματικότερη πολιτική για τα ε, απόβλητα συνδυάσεις με τρόπο επιτυχή η εισηγήτρια. Στην κυκλική οικονομία προϊόντα και εξαρτήματα αυτών θα πρέπει να στο δυνατόν ε, να έχουν τόσο δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να υπάρχει δυνατότητα και της, α, ε, της και της διάλυσης και επανα συναρμολόγησης ε, των προϊόντων ώστε να μπορούν να επισκευαστούν και να υπάρχει βέβαια η πιο αποτελεσματική οικολογικά ε, χρήση των προϊόντων και διάθεση του στην αγορά. Functional economy, λοιπόν, λειτουργική οικονομία με πολλά πλέον εκτήματα για μένα και ιδιαίτερα η γνωμοδότηση έχει μεγάλη σημασία γιατί απαντά στο ερώτημα πώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση ενός προϊόντων, Στο 2 η εισηγήτρια επισημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικά υποδείγματα χρήσης και κατανάλωσης στα υβριδικά προϊόντα. Εδώ λοιπόν θα έχω κάποιες επικρίσεις αγαπητοί συνάδελφοι. Τι μπορεί να είναι μια ε, γιατί πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική μια υβριδική λύση, εάν είναι ε, αποτελεσματικό το προϊόν που έχω, είναι καλής ποιότητας και δεν χρειάζεται να το αντικαταστήσω, ε, τότε είμαι καλυμμένη ως προς την διάρκεια ζωής, ως προς την εξοικονόμηση των πόρων και της ενέργειας και όλα αυτά. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει μια διαφορετική τεχνολογία να δώσει άλλες λύσεις. Εδώ θα ήθελα προς εξηγήσει λοιπόν. Ιδιαίτερα η ενίσχυση της αρχής ε, της ε, ευθύνης του παραγωγού που εισάγεται στην οδηγία πλαίσιο είναι θετική ε, για μένα. Πρέπει να έχουμε πιο έντονη εμπλοκή των παραγωγών με την έννοια της ευθύνης. Πολλά κράτη-μέλη έχουν δώσει ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερη σημασία την ε, παράταση τη ζωή των προϊόντων. Η Γαλλία έχει παραδείγματι καταστήσει ποινικό αδίκημα την εσκεμμένη συντόμευση ζωή, Η Νορβηγία προχωρεί σε αντίστοιχε ρυθμίσει. Το Βέλγιο προσπαθεί να εξασφαλίσει μέσω τη προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντο ε, τι σχετικέ εξελίξει. Στη Γερμανία είναι ανάγκη να υπάρχει μια αντίστοιχη ε, τάση. Και βέβαια η ε, οικολογική σήμανση από το 1978 ισχύει στη Γερμανία. Η ενίσχυση λοιπόν της μακροβιότητας των προϊόντων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Σε αυτό θα ήθελα να κάνω μια τροπολογία στη συνέχεια όταν είναι έτοιμο το κείμενο. Χρειάζεται ευρωπαϊκό συντονισμό ώστε να μην εισάγονται μεμονωμένε διατάξει που θα παρεμποδίσουν την απόσκοπτη λειτουργία τη ενιαίας αγορά. Και βέβαια αυτονόητο θα πρέπει να είναι να ε, προαχθεί η μεγαλύτερη διάρκεια ζωή των προϊόντων και η βιωσιμότητα, η αηφορία ταυτόχρονα με την ενίσχυση και της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η έκθεση πρωτοβουλίας μπορεί να εξισορροπήσει μεταξύ και της αηφορίας στην παραγωγή μέσα από μια κυκλική οικονομία και της εξασφάλισης ενός πεδίου καινοτομία χάρη σε νέα κίνητρα. Καλή βάση λοιπόν συνεργασίας και προσβλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρίση έχει το λόγο. Θα μιλήσω εξ ονόματος της κυρίας Μάισνερ που δεν μπορούσε να είναι παρούσα για την, στη συνεδρίαση αυτή η Γκεζίν. Καλωσορίζει την ε, έκθεση αυτή έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη το αποτύπωμα αυτό και τις παραμέτρους έτσι ώστε να ε, μην φτάνουμε σε απόβλητα και επίσης να υπάρχει τρόπος ε, μεγαλύτερης διάρκειας ζωής για τα προϊόντα και στη συνέχεια η απομάκρυνσή τους. Υπάρχουν οι πρώτες ύλες καταρχήν και ως προς την ε, απομάκρυνσή τους οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τις ε, κατάλληλες υποδομές για αυτό. Για αυτήν. Η Γκεζίν Μάισνερ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση σε σχέση με την ε, απομάκρυνση ε, αυτών των προϊόντων και δεν ξέρει κατά πόσο η τεχνολογία επιτρέπει την αποκατάσταση προϊόντων και σε αυτή την περίπτωση ποια θα ήταν η κοστολόγηση. Θα πρέπει να βρούμε μία σωστή εξισορρόπηση μεταξύ καινοτομίας και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, ιδιαίτερα στο σημείο 1α. Επίσης, η συμπεριφορά του καταναλωτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ε, επαγρύπνησης και συνειδητοποίησης και αυτό αφορά την αιτιολογική σκέψη α. Και συμφωνεί λοιπόν με την προσέγγιση του εισηγητή Τώρα, σε σχέση με την παράγραφο 4 θα ήθελα να πω εγώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για την ε, ε, οικολογική προσέγγιση του ζητήματος. Είχαμε συνεργαστεί με τους Λίζε και Τούρμες για μια προγενέστερη έκθεση και μιλήσαμε για μια πίεση έτσι ώστε να δράσουμε εξ αρχή σε σχέση με τον ε, κύκλο ζωής του προϊόντος γιατί έτσι μπορούμε να προβούμε σε ένα 80% ε, εξοικονόμησης. Γι' αυτό θεωρώ ότι για τους φιλελεύθερους η προθεσμία της παραγράφου 4 είναι υψίστης σημασίας. Ευχαριστούμε κυρία Ρίσ. Ε, ο κύριος ε, Χουαρίστη Αλόνς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δέχομαι την προσέγγιση του εισηγητή, αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε ε, ότι ο κύκλος ζωής θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ε, προϊόντων ήδη από το σχεδιασμό τους για να μην υφίστανται ευθορά γρήγορα και να υπάρχει η διαδικασία ε, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Και υπάρχει ένα σχεδιασμός μέχρι το 2019. Θα μπορούσε η Επιτροπή να μας πει τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έτσι ώστε να προβάλλουμε συγκεκριμένα πρότυπα κατασκευής ε, σεβόμενοι το περιβάλλον. Ως προς τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, πολλά μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε τον ε, κατάλογο νέων προϊόντων που ε, αφορά ένας, έναν κοινό σχεδιασμό. Επίσης θα πρέπει η βιομηχανία να απομακρυνθεί από αυτό το σχήμα κατασκευής, χρήσης και απομάκρυνσης ε, δηλαδή απόρριψης του προϊόντος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλή πρακτική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνεργασία των τοπικών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαδικασία επισκευής ή ανταλλαγής προϊόντων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο είναι πιο βιώσιμο που να βασίζεται σε, στη συνεργασία και όχι στον ατομισμό. Μιλάμε για μια καταναλωτική κοινωνία η οποία προβαίνει σε αποκλεισμούς. Ήδη από την παιδική ηλικία προβάλλεται αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο και οι τροπολογίες μας θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, και φυσικά θα έχουμε επικοδομητική προσέγγιση των δεδομένων της ε, εισήγησης. Παντιτσίνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια πρωτίστως. Θα θέλαμε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα προϊόντα και αυτό σχετίζεται με την πολιτισμική μας, με την πολιτισμική μας ε, προσέγγιση. Θα πρέπει όμως να δούμε ποιος είναι ο εχθρός. Αυτός ο, ο φιλελευθερισμός ε, δημιουργεί νέα προϊόντα, τα οποία όμως οδηγούνται σε απομάκρυνση στη συνέχεια. Δηλαδή, είμαστε και καταναλωτές, ζούμε σε μια κοινωνία του καναλωτισμού, όπου ο καθένας θέλει δύο πλυντήρια, δύο τηλεοράσεις και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε να υπάρχει υψηλότερος καταναλωτισμός. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πολλά χρόνια ζωής, αλλά δυστυχώς απομακρύνονται από την αγορά και αυτό απομακρύνει και τους βιοτέχνες. Έτσι μπαίνουν στην αγορά ολοένα και νεότερα προϊόντα τα οποία δείχνουν ότι τα προηγούμενα είναι παροχημένα, όπως ισχύει με τα κινητά μας. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για αυτή τη την προσέγγιση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λοιπόν τα προϊόντα και στο τέλος της ζωής τους θα πρέπει να αποσυναρμολογούνται και να ξαναχρησιμοποιούνται τα μέρη τους. Θεωρώ ότι έτσι θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και θα μειώσουμε τα απορρίμματα, τα απόβλητα. Ο παραγωγός έχει την πλήρη ευθύνη του προϊόντος έτσι ώστε να δημιουργούνται προϊόντα που να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορνάνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εργασία της όσον αφορά ε, την προκαθορισμένη διάρκεια ζωής. στις ε, αναπτυσσόμενες, στις ε, χώρες ε, βλέπουμε ότι έχουμε 468 κιλά απόβλητα ανά άτομο στις, στους δήμους και στις κοινότητές μας. Έχει αυξηθεί δηλαδή το βάρος των σκουπιδιών μας. Αυτή η προγραμματισμένη λοιπόν μείωση της ζωής των προϊόντων αποτελεί κατάχρηση ε, και μπορεί να ε, σημαίνει ε, οτιδήποτε για οποιοδήποτε προϊόν. Μπορεί να είναι το καλτσόν το οποίο βγάζει πόντους αμέσως ή ένα ηλεκτρικό, μια ηλεκτρική συσκευή η οποία δεν λειτουργεί παραπάνω από χήφορες. Στην Γαλλία υπάρχει σχετική νομοθεσία η οποία απαγορεύει την, τον περιορισμό της, ε, ε, της διάρκειας ζωής. Ωστόσο ε, γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχει βάση των αρχών του ανταγωνισμού ευρεία χρήση αυτής της ε, ε διάρκειας ζωής. Αυτό το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε θα είναι να αναφέρεται σαφώς η απαγορεύση και τις οδηγίες χρήσεως ε, των προϊόντων και βεβαίως το πρώτο βήμα θα πρέπει ε, να είναι να ε, εφαρμοστεί ο νόμος και όπως λέει και η συγγήτρια πολύ σημαντικό βασικό ε, στοιχείο και προϋπόθεση για την όλη διαδικασία είναι ο καταναλωτής να ευαισθητοποιηθεί. Δεν ε, θα πρέπει μονάχα οι επιχειρήσεις ε, να έχουν την ευθύνη. Θα πρέπει οπωσδήποτε και οι δημόσιες αρχές να προωθήσουν την σωστή και οικολογική χρήση των προϊόντων. Ε, ας πούμε, αναφερόμαστε εδώ ε, ενδεχομένως στο φιάσκο ε, των λαμπτήρων LED, τα οποία τώρα βρίσκονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και τα οποία με πολύ μεγάλες φανφάρες οι διάφοροι φορείς είχαν προωθήσει. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες στο κείμενο της εισηγητρίας που θα πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λίζε. Και ευχαριστώ τον κύριο Στυλ και, την κυρία Λάνιεν που παρουσίασε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα ήθελα να, να συμπληρώσω ακόμα ένα-δύο σημεία, υποστηρίζοντας βέβαια την έκθεση και τα σχόλια της κυρίας ε, Λάνιεν. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα θα σας ε, δώσω που θα πρέπει να μας απασχολήσουν πιστεύω Είναι βεβαίω πολύ θετικό το ότι έχουμε όλο και περισσότερα, περισσότερους λαμπτήρες LED. Ταυτόχρονα έχουμε πρόβλημα ως προς την ανάγκη αλλαγής του λαμπτήρα, εάν αυτός είναι σε λάθος χρώμα φερρυπίνη, εάν χαλάσει πρέπει να πετάξουμε ολόκληρο το μηχάνημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι σωστή επιλογή είναι περιορισμένα δηλαδή τα ανταλλακτικά στους λαμπτήρες LED που μπορούμε να αλλάξουμε. Επίσης, τα αγαπημένα μας smartphone. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όταν βγαίνει ένα νέο iPad στην αγορά, αρχίζει και αυξάνεται σιγά σιγά η καθυστέρηση στην λειτουργία Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό να κοιτάξουμε την δυνατότητα για διατήρηση των updates, της ενημέρωσης λογισμικού που προβλέπεται για παλαιότερα ε, μηχανήματα για παλαιότερες συσκευές, ώστε να μην χρειάζεται ο καταναλωτής να προβαίνει σε αγορά νέου ε, μηχανήματος κάθε τόσο. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η Επιτροπή. Ίσως υπάρχουν και άλλα επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία ε, έχουν μια τέτοια, τέτοια κατάσταση. Επίσης, δεν ξέρω αν μπορούν να αρκέσουν πάντα τα οικολογικά μέτρα στο να δώσουμε λύσεις. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε και εναλλακτικέ και η Φρεντερή Κρίση αυτό έχει δίκιο, ήταν και η συγγήτρια πριν από τόσα χρόνια, μια πολύ επιτυχημένη έκθεση, γιατί είχαμε πολλά καταφέρει σε σχέση με την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργεια. Ωστόσο, κάποια ζητήματα που παρέμεναν δύσκολα, που είχαν αρκετά προβλήματα, άφησαν μεγάλο πεδίο ανάπτυξη τη επιχειρηματολογία των πολεμίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν οικολογικό σχεδιασμός, ναι. Μπορούν να λυθούν όμως όλα τα προβλήματα με αυτόν. Όχι. Δεν είμαι τόσο σε βέβαιος τουλάχιστον εγώ. Και έτσι καλό θα ήταν να προτείνουμε από κοινού να καλλιεργηθούν και άλλες εναλλακτικέ στο δημόσιο διάλογο. Φιλιππίν, μια καλύτερη σήμανση όπως για το θέμα του λαπτήρα LED Πρέπει να υπάρχει σήμανση. Πολλές φορές υπάρχει, δεν ξέρουμε καν ο καταναλωτής τι διαβάζει, οπότε ίσως θα πρέπει να είναι καλύτερη η ανάρτησή της, ε, πιο ευανάγνωστη, πιο κατανοητή. Επίσης για ορισμένα προϊόντα θα μπορούσε να δοθεί παράταση εγγύησης υποχρεωτικά από τον νόμο. Όταν λοιπόν έχω μία ε, λάμπα, ένα λαμπτήρα, μία λάμπα τη οποία της οποίας δεν μπορώ να αντικαταστήσω, τότε ας παρατείνεται η διάρκεια ζωής η, η εγγύηση ως προς τη διάρκεια ζωής. Γιατί τότε, εάν τυχόν σταματήσει να φέγγει αυτός ο λαμπτήρας, θα πρέπει να αντικαταστήσει ολόκληρη τη λάμπα. Ας το καλύψουμε με την εγγύηση λοιπόν. Και θα ήθελα και η Επιτροπή να μας πει πού είναι ακριβώς το πρόβλημα σε αυτό. Εάν έχω ένα προϊόν το οποίο ε, σταματάει να δουλεύει νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, Πού είναι η προστασία του καταναλωτή, γιατί δεν κάνει κάτι, γιατί στη τελευταία ανάλυση ε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και μέσω των ανταγωνιστών. Πώς θα πέσει ένα προϊόν ε, στην αγορά συνέχεια το οποίο επιβαρύνει με μεγαλύτερο κόστος ε, κάθε εμπλεκόμενο και βέβαια πάνω από όλους τους καταναλωτές δεν υπάρχουν μέτρα να ληφθούν. Κλείνουμε λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Στρέλακ έχει το λόγο. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για, την αυτή, για το εξαιρετικό αυτό προσχέδιο γνωμοδότησης για τα μέτρα αυτά που εντάσσονται στην κυκλική οικονομία και νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση και με τις τροπολογίες μας. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο έχει σχέση με τον ε, οικοσχεδιασμό ε, που έχει μεγάλη σημασία με την βιομηχανία έτσι ώστε να έχουν ε, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τα προϊόντα αλλά και να μπορούν να επισκευαστούν γιατί αυτό θα δημιουργούσε και νέες θέσεις εργασίας και θα ενίσχυε τις τοπικές οικονομίες καθώς και να ενισχύσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας που έχει μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, γιατί με αυτή την προσέγγιση θα υπάρχουν περισσότεροι πόροι και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποδοτικοί και σε άλλες πολιτικές σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας. Υποστηρίζω λοιπόν την ε, μετάταξη των προϊόντων από προϊόντα σε υπηρεσίες, γιατί αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε νέα πρότυπα και ένα νέο επιμερισμό ε, ευθυνών στην οικονομία. Περνάμε λοιπόν από τα αγαθά στις υπηρεσίες, κάτι το οποίο συνεισφέρει στα κίνητρα προς την ε, βιομηχανία και τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τη ζήτηση, δηλαδή τα προϊόντα θα είναι ε, πιο δαπανηρά από ό,τι σήμερα, γιατί σήμερα δεν συμπεριλαμβάνεται το περιβαλλοντικό κόστος ε, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, συσκευές αυτές ε, ως προς συσκευές και προϊόντα. Γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση και πληροφόρηση των καταναλωτών. Γιατί δηλαδή είναι καλύτερη αυτή η προσέγγιση αγοράς προϊόντων που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά και είναι λίγο πιο δαπανηρά και γιατί ενισχύουμε την τοπική οικονομία με βάση τη ε, διαδικασία επισκευής αυτών των προϊόντων. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ενσυνειδητότητα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δοθούν οικονομικά κίνητρα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάλσο έχει το λόγο είναι ο τελευταίος ομιλητής. Κυρία... Ευχαριστώ πολύ. Ε, που μου δίνετε το λόγο. Ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θα ήθελα να σημειώσω δε το σημείο 6 ε, και το θέμα της ε, οικολογικής επισήμανσης. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει αγοράζοντας ένα προϊόν να ξέρουμε την διάρκεια ζωής του. Ο καταναλωτής ε, δεν θα πρέπει να ενθαρρύνεται να αγοράζει προϊόντα ε, προϊόντα τα οποία δεν, ε, για τα οποία μάλλον δεν διαθέτει πολλές πληροφορίες και τα οποία δεν ε, είναι βιώσιμα. Σε μερικές φορές ακούμε ας πούμε ακούμε διαφημίσεις αυτοκινήτων που λένε το αυτοκίνητο αυτό έχει διάρκεια ζωής ε, ε, μεγάλη, οτιδήποτε. Αλλά σε γενικές γραμμές ε, οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να αντικαταστήσουν τα προϊόντα, να αντικαθιστούν μάλλον τα προϊόντα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το σημείο αυτό της ημερησίας διατάξεως, γιατί κυρίως για κινητά τηλέφωνα, αυτά τα iPhone και τα περίεργα τηλέφωνα, ε, που κάνουν ιδιαίτερα επιθετική ε, πολιτική και ιδιαίτερα επιθετική διαφήμιση ε, έχουν σαν αποτέλεσμα ο καταναλωτής εύκολα να πετάει το προϊόν και να μην αντικαθιστά. Εγώ έχω, και το, σας το δείχνω στο χέρι μου, ένα τηλέφωνο Nokia το οποίο αγόρασα πριν από τρία χρόνια και τώρα πρέπει να το πετάξω γιατί δεν βρίσκω μπαταρία, δεν βρίσκω φορτιστή, ε, δεν έχω, δεν, δεν μπορώ να βρω φορτιστή πουθενά, σε κανένα μαγαζί. Όπου και να τον ζήτησα μου είπαν δεν πρόκειται να βρείτε τέτοιο φορτιστή, καλύτερα είναι να αγοράσετε ένα καινούριο τηλέφωνο, γιατί τέτοιο φορτιστή για αυτό το τηλέφωνο δεν πρόκειται να βρείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ε, και ε, η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πάμε, έχει κλείσει ο κατάλογος. Ο κύριος Μπένετ έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να σχολιάσετε. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπάρχουν ε, ορισμένα σημεία που θα πρέπει να τονιστούν. οι Επιτρόποι. ε, ε, συμφωνεί με πολλά από τα στοιχεία αυτής της γνωμοδότησης καθώς και με την αρχική γνωμοδότηση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτός ο οικολογικός ε, σχεδιασμός ε, λαμβάνει υπόψη το χαμηλότερο κόστος για τη διάρκεια ζωής, για μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, έτσι ώστε να συμβαδίσουμε και στην τιμολόγηση αυτών των προϊόντων. Γι' αυτό όταν μιλάμε για επισκευασιμότητα και νέα χρήση, εκ νέου χρήση, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αυτήν την ελαχιστοποιημένη προσέγγιση κόστους. Υποβλήθηκαν ορισμένες ερωτήσεις και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι μία από τις βασικές μας προκλήσεις. Χαμηλότερο κόστος με υψηλότερη διάρκεια ζωής. Τώρα, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης σε σχέση με την ανακυκλωσιμότητα και την επισκευασιμότητα. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι υπάρχουν 30 τεχνικές επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα αυτό και 7 ε, οριζόντιες ομάδες και μεταξύ 18, τελευταίο εξωμήνου 18 και πρώτου του 19 θα ε, μας αποδώσουν τους καρπούς της εργασίας τους. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν στοιχεία που είναι πιο οριζόντια από ό,τι άλλα και ως προς τις αντισταθμίσεις ανάλογα με την σπουδή και την τεποποίηση δέχτηκαν να έχουμε τρία είδη τεκμηρίωσης, τυποποίηση ΙΕΝ, υψηλότερη, τεχνικές προδιαγραφές και συμφωνίες εργαστηρίων ΣΕΝ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για προϊόντα τηλεπικοινωνιών καθώς και άλλων που εξελίσσονται γρήγορα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ολόκληρον αυτό τον οικολογικό σχεδιασμό μέσα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας που κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αμφίδρομη πορεία μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησεων όπως βλέπουμε και από τα workshops για τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ του χρόνου σας. Μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις ενδεχομένως. Είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά σε σχέση με ορισμένα μέτρα τα οποία ε, προτείνουμε τώρα, για τον ε, κανονισμό του οικολογικού σχεδιασμού προσπαθήσαμε να Υπάρχουν ορισμένες απαγορεύσεις σε σχέση με μη αναστρέψιμες ε, τεχνικές, έτσι ώστε ε, φυσικά να μην υπάρχει, και μια, να μην υπάρχει τόσο νομικίστικη προσέγγιση στο όλο ζήτημα και να μην υπάρχει ε, απόλυτη δέσμευση και φυσικά στις υπηρεσίες ως προς τα PC και άλλο ε, hardware που χρησιμοποιούμε, το θέμα αυτό έχει προωθηθεί. Το λογισμικό ή phoneware, όπως ορίζονται αυτές οι υπηρεσίες, δηλαδή το νέφος και ούτω καθεξής, ε, αφορά έναν δεύτερο κύκλο ζωής του προϊόντος και εδώ χρειάζεται το κατάλληλο λογισμικό. Ε, πρόκειται για αρχικά μέτρα που προσπαθούμε να προωθήσουμε και αυτό συμβαδίζει και με το λειτουργικό μέρος του προϊόντος, δηλαδή τους drivers και τα ε, ηλεκτρονικά, το ηλεκτρονικό σκέλος και εξαρτήματα θέλουμε να μειώσουμε την ποσότητα η οποία καταστρέφεται. Αυτό βεβαίως, δηλαδή η καταστροφή αφορά και ζητήματα απορρίτου και δεν μπορούμε ε, να αναγκάσουμε τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να μην καταστρέφουν αυτά τα στοιχεία των σκληρών, γιατί, των σκληρών δίσκων, διότι το θέμα του απορρίτου είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, σε σχέση δηλαδή με τα περιβαλλοντικά. Αλλά το θέμα της καταστροφής ε, των στοιχείων είναι ύψης της σημασίας, δηλαδή προσπαθούμε να υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος ζωής, πέρα από θέματα απορρίτου έτσι ώστε να υπάρχει και δυνατότητα καταστροφή στοιχείων που να διατίθενται εξ αρχής με το λογισμικό το οποίο αρχικά απολύται στον καταναλωτή. Έτσι θα είχαμε περισσότερες συσκευές για να προωθήσουμε ένα δεύτερο κύκλο ζωής τους. Εάν ε, θεωρείτε ότι δεν έχω απαντήσει, είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια όλους τους συναδέλφους. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι θα έχουμε μια εξαιρετική έκθεση ύστερα από αυτή τη συνεργασία. Θα σταθώ σε ένα-δύο σημεία μόνο. Στα όσα είπε ο κύριος Λίζε. Είναι σωστό αυτό που επισημαίνει Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε την ε, πρόκληση ε, των software που υπάρχουν σε παλαιότερα μηχανήματα, υπολογιστές κτλ. Για την κυρία Κόλλη θα συμφωνήσω στο θέμα των προβλημάτων που επισήμανε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να δώσουμε κάποια κίνητρα στην βιομηχανία για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων που θα παράγονται ώστε πραγματικά να φτάσουμε στην κυκλική οικονομία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, Μια πραγματική κυκλική οικονομία. Ένα σαφέ μήνυμα βεβαίω θα πρέπει να αποστολεί και ταυτόχρονα να μπορέσουμε χάρη και στο leasing να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη διάρκεια των προϊόντων. Ίσως αυτό να βοηθήσει ως... Ε, Ευχαριστώ πολύ. 8 Μαρτίου, προθεσμία για τις τροπολογίες 12 το μεσημέρι. Προχωρώ στο επόμενο θέμα ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμυνα στα τρόφιμα, τη σχετική με τρόφιμα και δίνω το λόγο στον Διευθυντή Ράιν, Γενική Διεύθυνση Υγείας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πω δύο λόγια εισαγωγικά για τις νομοθετικές ρυθμίσεις, το σύστημα ε, κινδύνου που έχουμε η ε, επισήμανσης κινδύνου. Ξεκινώ λοιπόν με την ε, νομοθεσία τη σχετική με την υγεία. Υπάρχει η σχετική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σοβαρούς διασυνοριακούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ενημερωνόμαστε λοιπόν και καταγράφονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων ε, με στόχο την αξιοποίηση στις αιτήσεις εκθέσεις ε, διαφοροί κίνδυνοι. Έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης μεταξύ των κρατών μελών για να ενημερωθούν, ε, να αλληλοενημερωθούν για διασυνοριακά προβλήματα αλλά και επιδημίες. Έχουμε ένα σύστημα κοινού, κοινής αξιολόγησης κινδύνου για τις μεταδοτικές νόσους και άλλους τύπους απειλές όπως βιοασφάλειας. Εκεί αξιοποιούμε την, τις επιστημονικές μας επιτροπές για την αξιολόγηση του κινδύνου και η, και η Επιτροπή Βέβαια και Ασφάλειας ε, έχει την αρμοδιότητα του στονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο των μέτρων όταν αυτά χρειάζονται λόγω απειλής για τη δημόσια υγεία προερχόμενης από διασυνοριακή προέλευση. Έχουμε γενική νομοθεσία τώρα για τα τρόφιμα του 2002 σε σχέση με τα τρόφιμα. Ανοιχνευσιμότητα λοιπόν πλήρης των τροφίμων ώστε να εντοπίζεται η επιχείρηση στην οποία έχει ε, διατεθεί τροφή, είτε ως τροφή είτε ως ζωοτροφή. Ε, η σχετική νομοθεσία πρόσφατα μάλιστα αναθεωρήθηκε. Κύριε ευθύνη για την ασφάλεια στις τροφές και τις ζωοτροφές ε, ανήκει στις επιχειρήσεις που καλούνται να προβαίνουν στην αξιολόγηση με βάση τις αρχές του σημείου ελέγχου κρίσιμων ε, ε, ευάλωτων σημείων. Έχουμε περί τις 3.000 ε, κοινοποίησεις από τα κράτη-μέλη με το σύστημα αυτό. Έχουμε τον κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους που προσφέρει ένα πλαίσιο ελέγχων από τα ίδια τα κράτη-μέλη για την επαλήθευση της στήρησης της νομοθεσίας της σχετικής με με τις ζωοτροφές, με την ε, υγεία των ζώων. Τώρα βρίσκεται στην διαδικασία προσαρμογής μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διασυνοριακή εποπτεία και στο, στο ενδοκινοτικό εμπόριο, ώστε να αντιμετωπίζονται οι απάτες σχετικές με τα τρόφιμα. Πολύ σύντομα λοιπόν θα ήθελα να πω για την νομοθεσία τη σχετική με την υγεία των ζώων, ότι έχουμε εναρμονισμένους κανόνες αρχικά. Τώρα αυτούς αντικαθιστά ένα πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για να αποφεύγονται είτε οι εσκεμμένες είτε οι τυχαίες ε, απειλές, συμπεριλαμβανομένων και των δύο απειλών. Οι μεταδοτικές επιζωοτίες ε, κοινοποιούνται, γίνεται ανάλυση πολύ γρήγορα μέσα σε ώρες από την εκδήλωση επιδημίας ε, μπορεί να κλείσει μια περιοχή εκεί όπου εκδηλώνεται δηλαδή η ε, νόσος ένα σύστημα σε πραγματικές, σε πραγματικές συνθήκες ε, ενημέρωσης για την εκδήλωση επιδημίας, ε, σύστημα τράπεζας εμβολίων, ε, υλικού αναφοράς, ομάδων κτηνιάτρων που μπορούν αμέσως να αναπτυχθούν για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα επιζωτιών, όπως επίσης και ομάδες που έχουν να κάνουν και συστήματα που αφορούν την υγεία των φυτών με ένα σύστημα καταγραφής ενδεχόμενων ε, επιδημιών σχετικών με την υγεία των φυτών. Υπηρεσίες, ε, παραδείγματι υπηρεσία για την πρόληψη των ε, της μετάδοσης των μεταδοτικών νόσων, υπηρεσία για την διατροφική ασφάλεια, ε, υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ποιότητας των τροφίμων ή των κινδύνων του ε, με παρακολούθηση των ε, κινδύνων που μπορεί να προκύπτουν με ένα σύστημα επαγρύπνησης και σε εγκάρσιο επίπεδο έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης στο CBRN που έχει να κάνει με βιολογικούς, χημικούς, πυρηνικούς και άλλους κινδύνους ε, σχετικούς με την ασφαλεία των τροφίμων ή τη δημόσια ειδικία που παρακολουθεί σε τακτική βάση με τις ε, εκθέσεις του αλλά και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη της εξελίξης και σε διεθνές επίπεδο κυρία Πρόεδρε. Έχουμε συνεργασία μεταξύ του Συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Υγείας ε, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και με όλους αυτούς τους συνδέσμους που προανέφερα. συνεργασία με την οργάνωση της Ατλαντικής Συμμαχίας ΝΑΤΟ για την δυνατότητα εντοπισμού ε, περιστατικών και ανείχνευσης του ταχύτατα, συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων, με πρώτη διάσκεψη για, τους για τη μείωση των βιολογικών κινδύνων στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2015, από την οποία προκύπτει μια σειρά από συστάσεις και αρκετές ε, άλλες οργανώσεις ή οργανισμούς με τους οποίους έχουμε τακτικά συνεργασία σε θέματα σχετικά με την προστασία της υγείας των τροφίμων, τη δημόσια υγεία και το καθεξής. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Σκαρσία. Σκαρσία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ε, Κομισιόν ε, για την παρουσία της για ένα θέμα όπως είναι αυτό της Food Defense που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας περιέγραψε η Κομασιόνα ε, την ε, νομοθεσία που έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή σχετικά με τα προϊόντα τα οποία φτάνουν στους καταναλωτές και που οπωσδήποτε είναι τα σιγουρότερα, τα ασφαλέστερα στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι γεγονός ότι εμείς έχουμε τις πιο, τους πιο αυστηρούς κανόνες στον κόσμο και επομένως η κατάσταση για τους καταναλωτές στην Ευρώπη και τους άλλους καταναλωτές των χωρών όταν ε, ε, καταναλώνουν τα προϊόντα μας ε, η κατάσταση είναι πολύ καλή. Εδώ όμω μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για τρομοκρατία. Μιλάμε για την δυνατότητα τα ευρωπαϊκά προϊόντα να είναι ε, ε, ε, να είναι επιστοποιημένα έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν υποστεί κάποια τρομοκρατική, κάποια αλλίωση είτε από εσκεμμένη τρομοκρατική επίθεση είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εγώ έχω υποβάλει διάφορα ερωτήματα και ε, μόνη αλλά και με άλλους συναδέλφους και η Κομισιόν ε, Γενικώ μας δίνει την αίσθηση ότι υπό τον πρόεδρο Γιούνκερ δεν έχει τόσο πολύ τη διάθεση ε, να παράγει νέα νομοθεσία. Βεβαίως ε, ε, μαθαίνουμε ότι ε, όλοι είναι υπέρ μιας νομοθεσίας συγκεκριμένης με την έννοια ότι ήδη υπάρχουν πρωτόκολλα προστασίας αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία. Και βέβαια από τη μία πλευρά ε, υπάρχουν ε, ε, κάποιες ειδικέ αρχές οι οποίες όμως αφορούν στην ουσία τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι προστασία του δημοσίου τομέα. Θέλουμε μία νομοθεσία η οποία θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, να σας πω ότι όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουμε και θα είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Να σας πω ότι η παραγωγή ε, ειδών διατροφής ε, και, που, και αυτοί που εξάγουν προϊόντα τους, πραγματικά, εάν είχαν στα χέρια τους μία νομοθεσία, θα βρίσκονταν σε πολύ καλύτερη θέση. Με, τις, ιδιωτικές, με τους ιδιωτικούς κανόνες έχουμε πρόβλημα. Ε, ε, όσον αφορά τα κατάλοιπα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτό, ε, παρότι υπάρχουν αποφάσεις της Κομισιόν. Έπρεπε να έχουμε ένα, ένα κείμενο, έναν κανόνα και ο κανόνας ήρθε και ήταν ο 14001. Και εγώ είχα ασχοληθεί με αυτό και πριν γίνω βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Εάν ε, έχουμε λοιπόν και για τη food defense όχι έναν κανόνα ISO όπως είχαμε πριν για τα κατάλοιπα ε, ε, αλλά ένα πραγματικό κανόνα ευρωπαϊκό τότε και οι εταιρείε, αλλά και οι καταναλωτές θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση. Δεν πρόκειται για μεγαλύτερη δαπάνη χρημάτων, αντιθέτως και αποταμίευση γίνεται και όλοι είναι πολύ πιο ήσυχοι. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι αυτό το θέμα, η πρόκληση της ε, food defense ε, είναι ακριβώς ε, η δυνατότητα καθορισμού της προστασίας των τροφίμων αλλά και ολόκληρου του αγρογεωργικού τομέα κατά βιολογικής, φυσικής μόλυνσης ή οποιασδήποτε άλλης απειλής που θα μπορούσε να αμαυρώσει και την την ε, ε, ασφάλεια του καταναλωτή αλλά και την εικόνα των ε, επιχειρήσεων. Έχει ήδη αναφερθεί ότι στα πλαίσια τρομοκρατικών ενεργειών ενέργειες κατά της ασφάλειας των τροφίμων είναι πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνες κυρίως όταν γνωρίζει κανείς ότι μας λείπουν αντιβιωτικά, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια βακτήρια τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και εναντίον των οποίων κανένα ε, τρόπο δράσης δεν έχουμε, με όλα αυτά τα στοιχεία κατανοούμε το έβρος του προβλήματος. Δεν υπάρχει ε, συνολική ε, νομοθετική αντιμετώπιση. Μόλις ακούσαμε ότι υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά δυστυχώς για την ώρα όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις δεν υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση αντίθετα με τις ΗΠΑ ή με κάποιες μεμονωμένες χώρες όπως η Γαλλία ας πούμε. Γιατί στην Γαλλία η έννοια του food defense περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Visi Pirate για την ε, ε, επαγρύπνηση ε, κατά της τρομοκρατίας και επομένως είναι απόλυτα σαφές ότι χρειάζεται προστασία και σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να πω στην Κομισιόν ότι δεν μου φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων μου φαίνεται ότι δεν έχει κινητοποιηθεί ιδιαίτερα πάνω στο θέμα αυτό, δεν έχει σκύψει πάνω από το πρόβλημα αυτό δηλαδή. Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι δράσεις δράσεις ε, τις οποίες έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων ε, θα ήταν στην καλύτερη θέση έτσι ώστε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ε, αυτού του προβλήματος. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται σήμερα για να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η Επιτροπή μας μιλάει για όλο το νομοθετικό πλέγμα που προβλέπεται στην υπόθεση αυτή για να αντιμετωπιστούν οι απειλές διασυνοριακού τύπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πρόκειται για πράγματα τα οποία ανησυχούν τους πολίτες. Τα συζητούν τους απασχολούν η βιοτρομοκρατία, η βιολογική τρομοκρατία, η βιολογική επιμόλυνση, η βιολογική κίνδυνη είναι ζητήματα πολύ ανησυχητικά. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι υπάρχει κίνδυνος που σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις μεταφοράς τροφίμων διαθαλάσσης. όπου διαρωτώμεθα πώς μπορούν όλοι αυτοί οι κανόνες που αναφέρατε να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τους πιθανούς κινδύνους. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφέστατα προγράμματα, ξεκάθαρη νομοθεσία για τον περιορισμό του κινδύνου της ε, επιμόλυνσης. Δεν το έχει αντιμετωπίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτώ λοιπόν, πώς φτάσαμε στην ανάγκη να αναπτύξουμε πρόγραμμα για την ασφάλεια των τροφίμων και την άμυνα για τα τρόφιμα. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει. Θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή γιατί. Ευχαριστώ. Πεντητσίνη. Ναι, πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο την ε, τρομοκρατία της σχετική με αλλά και τις απάτες. Θα θυμόμαστε βέβαια το λεγόμενο βιολογικό στάρι, την παραποιημένη λεγόμενη αυθεντική μοτσαρέλα από γάλα βουβάλας, ε, όλα τα ζητήματα τα σχετικά με ντομάτες και την κάρποκι μεθυλουλόζη, το ε466, που εμφανίστηκε, ανοιχνεύτηκε σε λεγόμενες νοπές γαρίδες. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν και σας τα αναφέρω ε, γιατί χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων για την αποφυγή και των απατών αλλά και την αποτροπή ενδεχομένων τρομοκρατικών επιθέσεων ε, μέσω της επιμόλυνσης τροφίμων. Μπορεί να είμαστε θέση να προστατεύσουμε τους ε, πολίτες μας αν δεν είμαστε μάλλον σε θέση να, προστατεύσουμε τους πολίτες μας εναντί τέτοιων είδων, είδων ε, απατών, πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε από πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Ας κοιτάξουμε λοιπόν, ας κάνουμε τις επενδύσεις που χρειάζονται για να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως για την ενίσχυση των συστημάτων σήμανσης, ελέγχου, προελεύσεως ε, των τροφίμων, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύξουμε και τη σχετική ανταλλαγή πληροφοριών, συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση των πιθανών επιθέσεων σε για λόγους τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, μερικές παρατηρήσεις μόνο για να απαντήσω. Όπως είπα, έχουμε ένα γερό πλέγμα νομοθετικό, ενισχύει η Επιτροπή μεριμνά, και αυτό είναι από τις αρμοδιότητες άλλωστε και της Επιτροπής, ε, από ε, Προστασία του καταναλωτή ε, σε σχέση με την τήρηση της νομοθεσίας. Μερινά λοιπόν για την τήρηση της νομοθεσίας γίνονται και έλεγχοι ε, επί τόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε τρίτες χώρες με τις σχετικές εκθέσεις αναφοράς πεπραγμένων που διαβάζονται και στα κράτη-μέλη. Το δεύτερο, σε σχέση με τα συστήματα ε, έγκαιρης προειδοποίησης, θα αντιληφθήκατε ότι αναφέρθηκα σε 5-6 διαφορετικά που ισχύουν ανάλογα με το νομοθέτημα από το οποίο εξαρτώνται. Μία από τις προτάσεις λοιπόν που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας καλύτερος σύνδεσμος, διασύνδεση μεταξύ αυτών των συστημάτων, ώστε η ε, ενημέρωση που μπορεί να προκύπτει να περνάει και στις υπηρεσίες για την υγεία των ζώων ή των φυτών και αντίστροφα ε, βιολογικοί κίνδυνοι που μπορεί να είναι και εσκεμμένοι επίσης θα καλυφθούν έτσι. Θέλουμε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα δηλαδή προειδοποίησης. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με την ε, Παρασκευή και τις ε, ασκήσεις ετοιμότητας που θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, με της υπηρεσίας μας βέβαια πάντα, με τις αρχές για την υγεία των τροφίμων και τη δημόσια υγεία, για την ασφαλεία των τροφίμων και την δημόσια υγεία, συνεργασία πάντα με τα κράτη-μέλη και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και ε, αυτό είναι κάτι το οποίο διαρκώς προάγουμε. Για την τρομοκρατία και την ασφάλεια παραπέμπω στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια με την πρώτη έκθεση για την υλοποίηση αυτού του θεματολογίου ιδιαίτερος 12 Οκτωβρίου του 2016 συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε, όπου μία από τις πτυχές που αναφέρονται είναι η υλοποίηση, η βελτίωση της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας της σχετικής με την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα και ιδιαίτερα θα επισημάνω εδώ δράσεις εν εξελίξη σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λεγόμενους ήπιους στόχους, δηλαδή τμήματα της κοινωνίας που μπορεί να είναι εργοστάσια ή αλυσίδες προμήθειας, φερρυπίν αλυσίδα προμήθειας τροφίμων, που δεν έχουν ε, τόσο καλή ε, προστασία σε όρους υλικούς, ενώ υπάρχει καλή νομοθεσία ή ε, προστασία που παρέχεται σε όρους υλικούς είναι περιορισμένη και άρα προσπαθούμε με, την, με τις προτάσεις μας να ενισχύσουμε την ε, ε, προστασία, την ανθεκτικότητα της αλυσίδας προμήθειας, των αλυσίδων αυτών προμήθειας σε κάθε επίπεδο. Και έτσι κοιτούμε, και το είδα αυτό σε μια χθεσινή συνεδρίαση, τη δυνατότητα εντοπίζοντα συγκεκριμένες δράσεις σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, να ενισχύσουμε την ε, ασφάλειά μας και την προστασία που παρέχουμε, ιδιαίτερα σχέση με τους ήπιους στόχους έναντι τρομοκρατικών απειλών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συμμετοχή στη συζήτηση και περνούμε στο επόμενό μας θέμα που είναι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απροστατμένη διαδικασία τροποποίησης του των ε, καταλόγων επιχειρήσεων του Καναδά από τις οποίες ε, επιτρέπεται τα κράτη-μέλη να εισάγουν προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση και ξαναδίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει την παρουσίαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Μιλάμε για τη νομική βάση για αυτό τον κατάλογο, τον κανονισμό 354 και εδώ μιλάμε για προϊόντα ε, ζωικής προέλευσης ε, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Στο άρθρο 12 παράγραφος 4 μιλάμε για την αναθεώρηση αυτού του καταλόγου. Οι εισαγωγές επιτρέπονται από εγκαταστάσεις που καταγράφονται σε αυτό τον ε, κατάλογο και αυτό εγγράφεται στην πιστοποίηση κατά την ε, εισαγωγή. Γίνονται έλεγχοι για να ξέρουμε ότι παρτίδες αυτές προέρχονται ακριβώς από, αυτές, από αυτούς τους καταλόγους. Προβλέπεται μία περίοδος 30 εργασίμων και σε αυτές τις 30 εργάσιμες, κατά τις, από αυτές τις 30, κατά τις 20 τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν να γίνει μία προσθήκη στον κατάλογο. Ε, σύμφωνα με την εκτινιατρική συμφωνία με τον Καναδά έχουμε μία αντιστήχηση κανόνων υγείας, ε, ιδιαίτερα για τον οπό ε, τα ψάρια και τα παράγωγα των ηχθείων έτσι ώστε ο Καναδάς να δεχτεί τα πρότυπα και προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ε, μιλάμε για αντιστήχηση προϊόντων. Αυτός ο πίνακας εγκαταστάσεων αφορά αυτή την εξισορρόπηση και θεωρήσαμε ότι αυτή η ισοδυναμία παρέχει εγγυήσεις και μία απλουστευμένη διαδικασία. Έχουμε και τις ίδιες διατάξεις με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά όταν γίνονται εξαγωγές προς τον Καναδά και ο Καναδάς εφαρμόζει την απλουστευμένη διαδικασία, την απλοποιημένη διαδικασία, δηλαδή μέσα σε ένα διήμερο επιτρέπει τις, στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξάγουν προς τον Καναδά. Αυτή η απλοποιημένη διαδικασία εγγράφεται στην προϋπάρχουσα συμφωνία Έγινε λοιπόν μία συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά στην Κοινή Επιτροπή και έγιναν συστάσεις. Τα κράτη-μέλη συμμετείχαν σε αυτή την ε, Επιτροπή Κοινής Διαχείρισης για να υπάρχει ένας απλουστευμένος κατάλογος που ε, παρουσιάστηκε στη Μόνιμη Επιτροπή για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, καθώς και τις προσμίξεις τροφίμων. Θα, μια, θα υπάρξει και μια εσωτερική απόφαση, έτσι ώστε η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ που ασχολείται με την ασφάλεια τροφίμων να πιστοποιήσει αυτές τις επιστολές. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα του Ευρωβουλευτή, για τις περιπτώσεις που μη επιλέξιμα προϊόντα εξαχθούν από αυτές τις εγκαταστάσεις, ο Τζον Ράιν απάντησε όταν μίλησε για τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων. Ε, γίνονται έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Σαντέ γίνονται έλεγχοι και στον Καναδά. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολεί κατά τη διαδικασία επαλήθευσης είναι η συμμόρφωση του Καναδά σε σχέση με τα προϊόντα αυτά τα οποία θα εξαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τους ελέγχους λοιπόν ασχολούμαστε με αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης η οποία γίνεται ακόμα πιο ενισχυμένη, ιδιαίτερα κατά τις εξαγωγές ε, βοήου κρέατος. Οι καναδικές αρχές όταν ε, ε, εξάγουν προϊόντα υποπροϊόντα κρέατος πληρούν τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά τις εισαγωγές αυτές να γίνονται έλεγχοι όχι μόνο το, της πιστοποίησης, αλλά και έλεγχη, κτηνιατρική έλεγχη πριν εισαχθεί το βόλιο κρέας στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ελπίζω να σας απάντησα, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Στάρις. Eh, <coughs> σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτά που μας είπε. Πρέπει να σας πω ότι είμαι σημείο επαφής και μόνο το σημείο επαφής ε, για την ε, διατροφική ασφάλεια ε, και παρακολουθώ συχνά επομένως τους ελέγχους που ο οργανισμός αυτός έχει κάνει στο παρελθόν όσον αφορά την χώρα του Καναδά. 13 έλεγχοι έγιναν στον Καναδά από το 2004 μέχρι και τώρα. Όμως, όμως, ε, δεν ε, αφορούσαν τον οπό κρέας ε, και το ψάρι και τις εισαγωγές. Για αυτά τα προϊόντα έγιναν μονάχα δύο έλεγχοι, το 2010 και ένας τελευταίος το 2014. Ακολούθησε δημοσίευση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο του 2015. Στο σύνολο λοιπόν πρόκειται για αποτελέσματα αρκετά ε, πρόσφατα και αυτά που διαβάζω στην ε, έκθεση αυτή δεν είναι τόσο καθησυχαστικά, δηλαδή δεν μου δίνουν ε, έτσι, μεγάλη ασφάλεια για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Βλέπω λοιπόν τον κατάλογο των εξαγωγέων για τον Καναδά και αναφέρεται ότι υπάρχουν ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί όσον όσον αφορά την ενημέρωση, επίσης όσον αφορά τα, το βόλιο κρέας. Ε, επίσης ε, υπάρχουν ισχυρές αντενδείξεις όσον αφορά την εξαγωγή, ε, την εξαγωγή κρέατος από άλογα ε, δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι 100 μέρες πριν την ε, ε, εξαγωγή τους είχε σταματήσει η οποιαδήποτε λήψη φαρμάκων από τα άλογα αυτά. Ε, η κτηριατρική υπηρεσία λοιπόν δεν έχει δώσει όλα τα στοιχεία τα οποία ε, έπρεπε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν βέβαια όλοι δέχτηκαν τα συμπεράσματα εκτός από μία χώρα η οποία εξέφρασε επιφυλάξεις ισχυρές. Ερωτώ, μπορούμε να δεχτούμε μέσω εκτελεστικής πράξης και επί τη βάση του άρθρου 12 του κανονισμού Μπορούμε να δεχτούμε, λέω, ε, να γίνονται αλλαγές ε, και να ε, γίνονται και παραχωρήσεις σχετικά με καταγραφή επιπλέον εγκαταστάσεων όταν γνωρίζουμε ότι η κτηνιατρική υπηρεσία έχει εκφράσει επιφυλάξεις και όταν γνωρίζουμε ότι η διαδικασία στα πλαίσια της νομοθέτησης ήταν διαφορετική. Δεύτερον, πριν από δύο εβδομάδες εγκρίναμε τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά. Ε, αλλά όσον αφορά την εισαγωγή κρέατος, ε, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση των ποσοστών ε, και για τα πουλερικά και για το χείριο και για το βόλιο κρέας. 12-15 φορές παραπάνω τόνοι θα μπορούν να εξάγονται από τον Καναδά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει αυτής της συμφωνίας. Οκ, okay, είναι μια συμφωνία και πρέπει να δεχτούμε τις αποφάσεις οι οποίες ψηφίστηκαν από μεγάλη πλειοψηφία, όπως είπα και προηγουμένως και το επαναλαμβάνω. Όμως βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, όπου οι ποσότητες κρέατος έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και μάλιστα ε, μια στιγμή ε, χρονική όπου γίνεται λόγος ε, για απλούστευση ε, όσον αφορά τον αριθμό των εγκαταστάσεων που ε, μπορούν να ε, ληφθούν υπόψη για τις εξαγωγές ε, από τον Καναδά προς την Ευρώπη για προϊόντα που κρέατος. Όσον αφορά τους ελέγχους λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο στον Καναδά οργανώνονται ε, ε, ξεχωριστά, να ελέγξουμε δηλαδή κατά πόσον ε, οργανώνονται ξεχωριστά οι παρτίδες κρέατος που προέρχεται από ζώα που έχουν υποστεί θεραπείες, έχουν πάρει ορμόνες και τα ζώα τα οποία δεν έχουν πάρει ορμόνες αυξητικές για την πάχυνση των ζώων. Εξού και η ερώτησή μου η προσέγγιση, ε, η απλουστευτική ε, όσον αφορά αυτούς τους ελέγχους και εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τον αριθμό των εγκαταστάσεων που μπορούν να εξάγουν βόλιο ή χείριο κρέας ή και πουλερικά αυτή η απόφαση απλούστευσης, ρωτώ, είναι σόφρον απόφαση λαμβάνοντας υπόψη ε, και τις ε, ε, αποφάσεις που πήραμε στα πλαίσια της συμφωνίας ΣΕΤΑ αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της κτηνιατρικής υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν όπως είπαμε τον Ιούνιο του 2015. Αυτή είναι η ερώτησή μου λοιπόν. Ήταν σόφρον αυτή η απόφαση απλούστευσης. Thank you. Um, first on, on Ευχαριστώ. Σε σχέση με τους ελέγχους που έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια από τις διάφορες υπηρεσίες με αυτή δεν αναφέρθηκε μια... Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη μια, ε, έκθεση, ε, μια έκθεση ελέγχου που ήταν σχετική με την έκθεση του 2016. Αυτή δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Πάντως θα υπάρχει σαφέστατη παρακολούθηση από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με ένα πρόγραμμα δράσης που απαιτείται, αλλά και όχι μόνο πρόγραμμα δράσης. Γιατί δεν ε, το αρχαιοθετούμε το πρόγραμμα δράσης, υπάρχει και η παρακολούθηση της συνέχειας, τι συνέχεια δόθηκε. Για να μην λησμονούμε την ανάληψη δράσεων αναλόγως των ευρημάτων, αποστολές, έλεγχοι μετά τον Καναδά, ε, που θα γίνουν κατά την παραβολή με το τα δράσεως και ε, με επαλήθευση ότι αυτά τηρούνται. Και γι' αυτό νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα να συζητηθεί το νέο πρόγραμμα των ελέγχων, αυτοί θα στηρίζονται και σε διάγνωση κινδύνου. Φερρυπίν, πόσες ε, ταχείες ε, ε, κρούσεις του κόδωρα κινδύνου θα έχουμε, πόσα θύματα επαγρύπνησης, αναλόγως θα γίνουν και οι έλεγχοι. Ποσοστώσεις. Αν θέλετε. Ναι, λοιπόν, το δεύτερο, σχετικό με τις ποσοστώσεις. Και αυτό βεβαίω ήταν ε, μέσα στη συμφωνία. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις εξαγωγές. Ο κατάλογος δηλαδή έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις τις ευρωπαϊκές που τηρούν οι καναδικές επιχειρήσεις για να δικαιούνται να εξάγουν. Δεν επεκτείνεται ο κατάλογος. Δεν επηρεάζεται δηλαδή σε σχέση με τις ποσοστώσεις της Συμφωνίας ΣΕΤΑ. want Πρόεδρε, όχι, θα απαντήσω όμω εδώ, γιατί ζήτησα από τον κύριο Φαντέκ ε, ενημέρωση. Μα δεν σα έδωσα το λόγο, κύριε συνάδελφε. Στον κύριο Καπούτο είχα δώσει το λόγο. Α, με συγχωρείτε, λέει κύριο Στα, κύριο Καπούτο, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, δύο λόγια κάπω πιο γενικά μια και είναι εδώ η Επιτροπή. Η αξιολόγηση των ποιοτικών προδιαγραφών των τροφίμων από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν μπορεί να περιορίζεται σε έναν απλό τυπικό έλεγχο. Αν κάνουμε μια ευάθυνση λοιπόν στην αξιολόγηση πέραν των ελάχιστων μικροβιολογικών αναλύσεων και κάνουμε μια ανάλυση της πραγματικής ποιότητας των προϊόντων από τα εις πρώτες ύλες μέχρι την τελική διαδικασία παραγωγής θα βλέπαμε ότι οι προδιαγραφές ποιότητας της παραγωγής του Καναδά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ισότιμη με αυτή της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ο Καναδάς όσον αφορά τα προϊόντα ε, τα ευαλείωτα όπως ε, το κρέας σε παραδείγματι έχει ακολουθήσει παραγωγή με προδιαγραφές χρήσεως ακόμη και ορμονών ή άλλες διαδικασίες που μπορεί να είναι και επικίνδυνες με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και ναι, μπορεί τυπικά να ακολουθούν ε, τα HCCP και όλες τις άλλες προδιαγραφές υγείας, τις τυπικές προδιαγραφές οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να, εισαγάγουν στην να εξαγάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό αρκεί και καλύπτει τις ε, προδιαγραφές μας. Όπως και με την ΣΕΤΑ δηλαδή υπάρχει κίνδυνος στις καναδικές ε, επιχειρήσεις να προσφέρουμε ε, μια ελευκό επιταγή εις βάρος βεβαίως των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μια δυνατότητα εισαγωγής προς την Ευρώπη χωρίς να τηρούν τους όρους ε, επεξεργασίας ε, φυτοϊγιεινής, μη, μη γονιδιακά τροποποιημένων οργανισμών και όλα αυτά, τα οποία θα είναι εις βάρος ευρωπαϊκής αγοράς και δημόσιας υγείας. Και με εντυπωσιάζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να κάνει περαιτέρω ελέγχους δεν δηλαδή αναλαμβάνει το ρόλο της ως θεματοφύλακα αυτών των αρχών και των συνθήκων και της νομοθεσίας. Και επίσης μια νομοθεσία που βλέπουμε έκπληξή μου ότι είναι απλουστευμένη, ε, μια νομοθεσία δηλαδή για την αδειοδότηση, στην οποία θα έπρεπε να γίνεται διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και ορμόνε αφενό και λοιπόν επιχειρήσεων αφετέρου. Ενώ δεν ενημερώνεται ο καταναλωτή για την ποιότητα προϊόντων που θα βάλει στο τραπέζι του και που θα καταναλώσει. Κύριε Μαγκίνες. Πρόεδρε, ένα θέμα που ήγηρε ο κύριος Στάς για το ε, κρέας αλόγου που δεν έδωσε απάντηση η Επιτροπή και θέλουμε να γνωρίζουμε πώς είναι το έλεγχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κρέας αλόγου, για την εισαγωγή του στην διατροφική αλυσίδα σε σχέση με κανόνες που ισχύουν στον Καναδά και είναι διαφορετική. Θέλω απάντηση. Αν δεν έχετε τώρα πληροφορίες, να μας τις στείλετε γραπτός, γιατί θέλουμε τις ε, απαντήσεις. Ερχόνται σε επαφή μαζί μας ε, πολλοί στις ε, πατρίδες μας, στις εκλογικές μας περιφέρειες και θέλουμε να ξέρουμε τι είδους σωτημία υπάρχει. Κύριε Στά, σας έδωσα το λόγο για μία φορά. Εντάχει σας παρακαλώ. Ναι, ναι, εντάχει πράγμα. Πράγματι, Θα ήθελα να σας πω ότι σας ε, κοιτούσα, αλλά προηγήθηκε ο κύριος Καπούτο. Αυτός προσέλκυσε την προσοχή σας. Λέμε λοιπόν Ε, ότι αυτή η έκθεση καταρτίστηκε το 2015. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κατά πόσο θα δοθεί μία συνέχεια. όπως έγινε και με τις προγενέστερες ε, εκθέσεις του Ιουνίου Έφνης του 2015. Γιατί μιλάμε για έναν τύπο ελέγχου στον Καναδά, αλλά δεν δημοσιεύθηκε κάτι μετά τις νέες αποκαλύψεις που έγιναν. Γίνεται λόγος για μια νέα ποσόστοση η οποία ορίζεται από τη ΣΕΤΑ που δεν έχει καμία σχέση με τους ελέγχους ή ορίζει νέους οργανισμούς, νέους ελεγκτικούς οργανισμούς. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο απλουστεύονται οι διαδικασίες για να έχουν περισσότεροι οργανισμοί έλεγχο, γιατί αν θέλουμε να αυξηθεί η εξαγωγική δυνατότητα του Καναδά, μας ενδιαφέρει να υπάρχει και σωστός έλεγχος από τη δική μας πλευρά. Βαντάικ. Έχετε κύριε Βαντάικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρώτα. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ποιότητας, επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει και η Κομισιόν εδώ και πολλές φορές. Δηλαδή μιλάμε για συμφωνίες, δεν με τον δικό μας πύχη προδιαγραφών. Υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ Καναδά και Ήμων, αλλά ε, ακόμα και πριν γίνει συμφωνία δεν δεχόμασταν ε, την περίπτωση ε, συγκεκριμένων, εξαγωγής συγκεκριμένων κρεάτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μας. Γι' αυτό, αυτό ορίζεται και μέσα στα πλαίσια ε, ε, υπάρχει μέσα στην συμφωνία με τον Καναδά, αλλά φυσικά εκεί που γίνονται, γίνεται χρήση ορμονών δεν επιτρέπονται οι εξαγωγές. Σε σχέση με το κρέας αλόγου, όπως ξέρετε, ε, δόθηκε μία απάντηση από την Διεύθυνση ΕΦΚΟ και η όλη διαδικασία παρακολουθείτε για να αυξηθούν οι έλεγχοι σε σχέση με τα άλογα που θα σφαγούν και μετά θα αποσταλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να βρίσκονται για έξι μήνες υπό τον έλεγχο των καναδικών αρχών πριν γίνει η σφαγή. Υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις αγωγές κρέατος ε, από άλογο. Σε σχέση με τα προγράμματα δράσης, ε, τα στοιχεία της ΕΦΚΟ είναι διαθέσιμα καθώς και τα σχέδια ή προγράμματα δράσης τα οποία ε, υπάρχουν στην ε, ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Τώρα Πάμε στο τελευταίο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης. Εδώ πρόκειται για μία ανταλλαγή απόψεων που οργανώθηκε σήμερα, διότι σήμερα γιορτάζουμε ε, την Παγκόσμια ημέρα σπανίων νόσων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους πολιτές σε εκείνους που πλήττονται από σπάνιες ασθένειες και όπως ξέρετε η επίπτωση αυτών των σπανίων νόσων είναι πολύ μεγάλη και για τους ασθενείς και για την οικογένειά τους. Πολλές φορές δεν υπάρχει κατάλληλη πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει κατακαιρματισμός γνώσεων γιατί μιλάμε για μικρό αριθμό ασθενών και ε, γι' αυτό δεν υπάρχει και ανάληψη καθηκόντων ή δράσης. Τώρα θέλουμε, τη σημερινή ημέρα θέλουμε το κοινό να γνωρίζει την ύπαρξη των, των σπανίων νόσων και της ημέρας αυτής για τις σπάνιες νόσους και θα θέλαμε και οι φαρμακοβιομηχανίες, ε, οι επιστήμονες, και τα κλινικά πειράματα να συνεχίσουν να υπάρχουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι σπάνιες ασθένειες. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Γενικό Διευθυντή και θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο έτσι ώστε να αναφερθώ στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις ε, σπάνιες ασθένειες. Υπάρχει ένας κανονισμός ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ασχολείται ακριβώς με την ανάπτυξη φαρμάκων για, τας, για τις σπάνιες νόσους που έχει διευρυνθεί και από την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια συνολική προσέγγιση στο θέμα το, της, διάστασης δημόσιας υγείας που έχουν οι σπάνιες ε, ασθένειες. Εκεί συνιστώνται και δράσεις ε, σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, για τις ε, σπάνιες ασθένειες. αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο αφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις σπάνιες ασθένειες και εντός του πλαισίου αυτού αναφέρονται και διάφορα επιπλέον μέτρα όσον αφορά τον ρόλο των ε, εμπλεκομένων φορέων. Ε, πρέπει εδώ να σημειώσω ιδιαίτερο το ρόλο των μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων και των ενώσεων για τις σπάνιες νόσους ε, πρόκειται για, ε, για για μια οργάνωση ε, η οποία έχει 60.000 μέλη και αφορά 4.000 καλύπτει, 4.000 σπάνιες ασθένειες. Επίσης, στην υπηρεσία φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ομάδες εργασίας γιατρών που ασχολούνται ιδιαίτερως με τις νόσους, σπάνιες νόσους των παιδιών και ε, λαμβάνονται μέτρα για να ανακουφιστούν ε, αυτοί οι οποίοι πάσχουν από τέτοιες ε, σπάνιες ασθένειες. Βεβαίως το σημαντικό είναι η γνώση και η επιτήρηση του πεδίου. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν μητρώα των σπανίων ασθενειών. Εμείς έχουμε μεταφέρει κάποια από τα δίκτυα επιτήρησής μας και σε τις ε, ομάδες οι οποίες αφορούν ε, τις ε, γενετικές ανομαλίες, συγγενείς ανομαλίες και τα μητρώα των σπανίων ασθενειών. Έχουμε κοινή δράση υπό το πρόγραμμα ε, ε, HELT που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 που έχει ε, σχεδιαστεί ακριβώς έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η δράση που έχει προκύψει από τις ομάδες του Συμβουλίου ε, στα πλαίσια ε, αυτής ε, της κίνησης έρχονται σε επαφή διάφορες εθνικές αρχές έτσι ώστε η πληροφόρηση να είναι σωστή και έγκαιρη όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες και σε διοικητικό και σε ιατρικό επίπεδο. Επίσης έχουμε ένα κοινό και συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα έτσι ώστε ε, ε, ο τομέας της υγείας, η κοινότητα της υγείας ε, και η ερευνητική κοινότητα να έρθουν κοντά. Έχουμε εδώ ένα ισχυρό επίπεδο συγχρηματοδότηση που φτάνει στο 70% και αφορά πενταετή περίοδο. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική δέσμευση. Επίσης έχουμε δεσμευτεί σε πρόγραμμα για την καλύτερη ενημέρωση ε, και ευαισθητοποίηση για τις ε, σπάνιες νόσου Όσον αφορά την πρόσβαση ε, στην θεραπεία, γιατί αυτό αποτελεί προβληματισμό όλων των ασθενών και των οικογενειών του. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει συζητήσεις όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών ε, ε, σε θεραπευτικές ε, διαδικασίες και προς αυτή την κατεύθυνση τον Ιούνιο της προηγούμενης χρονιάς εγκρίθηκε μία πρόταση για πιο ισορροπημένη προσέγγιση στο θέμα των φαρμάκων και των φαρμακευτικών αγωγών η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα ε, στις νέες φαρμακολογικές εξελίξεις ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης ε, πρέπει να πω ότι έχουμε αναγνωρίσει από πλευρά της Κομισιόν ότι είναι πρόκληση η υψηλή τιμή, το υψηλό κόστος πολλών φαρμακευτικών σκευασμάτων και ε, πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει ε, να υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτό άλλωστε είναι και το συμπέρασμα της ομάδας STAMP που αφορά την αξιολόγηση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα. Πρέπει να βελτιωθούν οπωσδήποτε οι θεραπείες που προτείνονται. Πρέπει να πω ότι έχουμε δώσει ε, ε, παραπάνω από 129 φάρμακα τα τελευταία χρόνια και πάνω από 1035 αδειοδοτήσεις. Η Κομισιόν επίσης ε, ελέγχει το φαρμακολογικό νομοθετικό, φαρμακευτικό νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να δώσει χώρο στις πραγματικά καινοτόμες θεραπείες. Υπάρχει επίσης ένα πιλωτικό ε, ε, πρόγραμμα ε, με χρηματοδότηση από πόρους που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορά ακριβώς τις σπάνιες ασθένειες. Στόχος του προγράμματος είναι να δοθούν νέα, πιο αποτελεσματικά σενάρια για την αντιμετώπιση των σπανίων ασθενειών από, το 2000, από τώρα μέχρι το 2020. Σαν συνέχεια του προγράμματος που ολοκληρώνεται το 2017. Τέλος, European Reference Network. Αυτό ε, αυτό ε, δημιουργήθηκε ε, μέσω της οδηγίας για την φαρμακευτική διασταύρωση και την διασταύρωση, τη διασταύρωση των, της υγείας. Ε, σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μεγάλη αναφορά ε, στις ε, σπάνιες ασθένειες και με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε χώρες οι οποίες είναι πιο προχωρημένες να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες και εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Έξι είναι οι ομιλητές. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να προσθεθεί το όνομά του στον κατάλογο. Όχι. Ωραία. Κλείνει ο κατάλογος μιλητών Ο κύριος Λίζε είναι ο πρώτος. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καταπολέμηση των Σπάνιο νόσων και η στήριξη προς τους ασθενείς που πάσουν από σπάνιες νόσους είναι προφανώς καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις ε, χαμηλή συχνότητα αυτών των ε, νόσων και άρα είναι δύσκολο για την επιστήμη να βρει λύσεις, ε, να κάνει διαγνώσεις ακόμα αλλά και φάρμακα να δώσει και γι' αυτό δεν μπορεί ένα μεμονωμένο κράτος μόνο του να αντιμετωπίσει τις ανάγκες, να έχει ειδικού κτλ. Η Μόρμπους Κοσέ που έχει που πλήττει τον μεταβολισμό είναι μια σπάνια νόσος, τη γνωρίζω πολύ καλά για λόγους προσωπικούς και νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε συνεργασία για την καταπολέμησή της. Η Φωνσουάς Κώστατ είχε μια σχετική έκθεση. Νομίζω τώρα η ε, έκθεση πρωτοβουλίας να μετατραπεί σε νομοθεσία για να ενισχύσουμε την, την ανάπτυξη φαρμακευτικών μέσων, φαρμάκων και γενικά την ιατροφαρμακευτική ε, κάλυψη των ασθενών που πάσχουν από σπάνιες νόσους. Επίσης, προβλήματα βλέπω πολλές φορές σε σχέση με την υλοποίηση Θέλω ιδιαίτερα να το επισημάνω αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με χαρά άκουσα αυτό που μας είπε ότι θα υπάρχουν ε, πολύ σύντομα πλαίσια αναφοράς, δίκτυα αναφοράς στη διάθεση του κοινού. Πολύ καλό αυτό. Αλλά από την άλλη δικές μου πληροφορίες μου λένε ότι είναι κάπως Ε, ασταθές το σύστημα. Εάν θέλει ένας ασθενής που πάσχει από σπάνια νόσο να ε, μεταβεί σε άλλη χώρα στην οποία μπορεί να έχει την κατάλληλη αγωγή, να τύχει της κατάλληλης αγωγής, δεν υπάρχει πάντα η σχετική ευχέρεια. Ας μας δείξει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορεί να δώσει λύσεις για τους ε, ασθενείς πάνω απ' όλα που χρειάζονται να πάνε σε ένα άλλο κράτος. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και καταρχάς θέλω να εκφράσω ιδιαίτερα την ικανοποίησή μου για τις προόδους ε, για τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα, για τα οποία όντως είχα την εισήγηση πριν από ένα διάστημα. 17 χρόνια συγκεκριμένα ε, είχε περάσει σχετική έκθεση, έγινε δεκτή με πολύ θετικά σχόλια από όλους τους εμπλεκόμενους, ασθενείς, γιατρούς, φαρμακευτικά εργαστήρια και παρά τις οποίες επικρίσεις ή και αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπενθυμίσει ότι 129 ε, φάρμακα αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση θεραπεία των σπάνιων ασθενειών χάρη στον κανονισμό αυτών. Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν γιατί είναι πολλές ακόμη σπάνιες ασθενειές που όχι μόνο δεν έχουν ε, θεραπεία κατάλληλα η αγωγή αλλά ούτε μπορούν να διαγνωστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ιδιαίτερα το 10, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων για την καταπολέμηση των σπάνιων νόσων έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και θέλω να τη χαιρετήσω εδώ. Η Προεδρία της Μάλτας τώρα αποφασίζει να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα για το εξάμεινό της στις σπάνιες νόσους και του συγχαίρω. Γι' αυτό είναι εξαιρετική επιλογή. Γιατί, γιατί χρειάζεται να δώσουμε μια νέα όθηση στην καταπολέμηση των σπάνιων νόσων και με βάση βέβαια τις εξελίξεις επιστήμης και τις εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αναφορά στο ευρωπαϊκό, τα νέα μέσα και τεχνολογικής ακόμη ε, και τεχνολογίες αλλά και ενημέρωσης που έχουμε, η ανάπτυξη νέων αγωγών απαιτεί να προβούμε κι εμείς σε ένα νέο βήμα. Η ενισχυμένη συνεργασία λοιπόν μεταξύ των κρατών μελών και μόνο αυτή μπορεί να επιτρέψει την προσέγγιση και στην έρευνα και στην αγωγή την ε, τυποποίηση της αγωγής ή ε, άλλης φροντίδας και της ε, προσέγγισης στον ασθενή. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στην έκκληση της Προεδρίας της Μάλτας για την υλοποίηση αυτής της εντολής. Καθυστερούμε όμως και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα ως προς την έγκριση και διάθεση στην αγορά των φαρμάκων αυτών, αλλά και ως προς τον προσδορισμό των τιμών και βέβαια των συστημάτων αποζημίωσης στα κράτη-μέλη. Οι εθνικές αρχές πολλές φορές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμακευτικών αυτών προϊόντων, που εντωμεταξύ όμως έχει εγκρίνει η υπηρεσία φαρμάκων. Και αυτό σημαίνει και περισσότερε διαδικασίε και επανάληψη των αναλύσεων και εν τέλει καθυστέρηση για την πρόσβαση στην αγορά καινοτόμων ε, αγωγών που απολύτως χρειάζονται από τα ΟΗ, οι οποίες απολύτως εξαρτάται ο ασθενής που νοσεί από σπάνια νόσο. Μαθαίνω μάλιστα πρόσφατα ε, ότι υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που χρειάζεται να φύγουν, Ευρωπαίοι, χρειάζεται να φύγουν, να πάνε στις Ηνωμένε Πολιτείες, με μικρά παιδιά πολλές φορές και δύο και τρία στην ίδια οικογένεια, ε, σε πολύ μικρή ηλικία, γιατί πάσχουν από τόσο σπάνια νόσο που δυστυχώς είναι και άγνωστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα η διάγνωσή της δεν είναι δυνατή, για την οποία χρειάζεται πολύ δαπανηρή θεραπεία και αγωγή στις Ηνωμένε Πολιτείες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια οικογένεια που πρέπει να σταματήσει ακόμα και να δουλεύει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μετακομίσει για να ε, συνοδεύσει τα παιδιά της στις Ηνωμένε Πολιτείες. Καταλαβαίνετε τι κόστος συνεπάγεται αυτό για τις ευρωπαϊκές οικογένειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να δείξει ελεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους για τις σπάνιες ε, ασθένειες και επίσης είναι κρίμα. Έχουμε διεθνούς κύρους ε, εμπειρογνώμονες στην υπηρεσία. Οι εθνικές αρχές λοιπόν έρχονται να αμφισβητήσουν αποφάσεις της, φαρμακευτικής, της υπηρεσίας φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βάλει και το κύρος της αίμα αλλά και την αξιοπιστία της νομοθεσίας των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του κεντρικά οργανωμένου συστήματος εις βάρος της δημόσιας υγείας με συνέπειες σημαντικές καθυστερήσεις και στην χορήγηση αγωγής και βέβαια για τους ασθενείς ε, την υποχρέωση να αναζητήσουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση λύσεις και αγωγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τι σκοπεύει να κάνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Χάρη στην ε, Προεδρία της Μάλτας έχει ευκαιρίες Ας προχωρήσει λοιπόν και ας τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των ε, κανονιστικών τους αρμοδιοτήτων τα κράτη-μέλη, τηρώντας την νομοθεσία. Ιδάλλως πώς θα προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή και ταλαιπωρούμε τους ασθενείς αυτούς που πάσχουν από μια σπάνια ασθένεια. Έτσι. Δηλαδή είναι σπάνια, δύσκολο να βρεθεί αγωγή και ταυτόχρονα δεν τους, επιτρέψουμε, δεν τους επιτρέπουμε την πρόσβαση σε μια αγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια διπλή καταδίκη. Δεν επιτρέπεται στον 21ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Νταλή. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ράιεν για την παρουσία του και για τη συζήτηση αυτού του σοβαρού ζητήματος. Συμφωνώ και επαυξάνω αυτά που είπαν η Λίζε Γκροστέτ γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας για να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία ως προς κέντρα αριστείας, ιδιαίτερα στο τομέα των σπανίων νόσων. Και θα ήθελα να τονίσω αυτό που ανέφερε ε, ο κύριος Λίζε. Εγώ προέρχομαι από τη Μάλτα, είναι ένα μικρό κράτος και έχουμε μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την πρόσβαση σε καινοτόμα φαρμακοσκευάσματα γιατί πρόκειται για μία αγορά που δεν είναι δελεαστική, δεν είναι οικονομία κλίμακας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα και ιδιαίτερα εκείνες τις οικογένειες που έχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν σπάνιες ασθένειες. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει κατά το δυνατόν γιατί υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός διάθεσης σπόρων και πιστεύω ότι η κοινή δράση θα βοηθήσει και τους ασθενείς και τους εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Ράιεν μίλησε για πρωτοβουλίες των κρατών μελών, αλλά θα ήθελα η Επιτροπή να μεριμνήσει περαιτέρω για αυτά τα μέτρα, έτσι ώστε και τα μικρά κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση. πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ε, διασυνοριακή συνεργασία και το συντονισμό. Αναφέρθηκε και η έρευνα. Από το 2000 και ε, μετά έχουμε ε, προωθήσει 620 εκατομμύρια για τις σπάνιες νόσους, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την περαιτέρω έρευνα στις σπάνιες νόσους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα. Επίσης, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την κατάσταση για τους ασθενείς για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα που είναι διαθέσιμοι σε άλλα, σε κρατη κράτη-μέλη. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Επειδή ζήτησα να ενταχθεί αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τους συντονιστές και εσάς, Πρόεδρε. Για τα εισαγωγικά σας σχόλια θα πρέπει όσοι πάσχουν από σπάνιες ασθένειες να γνωρίζουν ότι μας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Όταν παρευρέθηκα σε μία συνάντηση η οποία έφερε τον τίτλο «Μην προωθήσετε το Brexit για ασθενείς ε, σπανίων νόσων». Θα ήθελα να πω ότι αυτό το ζήτημα με όθησε να ε, ζητήσω να ενταχθεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών έχει σώσει ζωές και με την συνεργασία γιατρών, ερευνητών και ούτω καθεξής έτσι ώστε να μεταβούν οι ασθενείς στις χώρες που διαθέτουν αυτά τα φάρμακα. Πολύ φοβούμαι ότι με το Brexit θα συρρυκνωθεί αυτή η δραστηριότητα γιατί ελέγχθη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγάλη πείρα σε αυτό το τομέα και μια μεγάλη κληρονομιά. Και αυτό ενισχύθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για ε, Brexit, ε, ολιστικά θα πρέπει να το δούμε και στις επιμέρους του πτυχές. Υπάρχουν επιπτώσεις που θα ήταν ολέθριες για τη δημόσια υγεία. Ξέρω ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να το σχολιάσει, αλλά εμένα με απασχολεί πώς μπορεί να επιδράσει το Brexit στην υγεία των πολιτών που πάσχουν από μια σπάνια νόσο. Επίσης, ε, ως προς την πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Γκροστέτ και στις αρχές του επόμενου έτους θα υποβληθεί μια έκθεση πρόοδου. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα προωθήσει η Επιτροπή την αναθεώρηση έτσι ώστε να προσελκύσουμε τα φαρμακοσκευάσματα που χρειάζονται για τις σπάνιες νόσους. ως προς την ε, προσβασιμότητα στη θεραπεία και την τιμολόγηση των σκευασμάτων θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτά τα απαραίτητα και άκρος δαπανηρά φάρμακα. Θα πρέπει όμως η Επιτροπή μας να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με τις σπάνιες νόσους. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που βάλατε το θέμα αυτό σε ημερήσια διάταξη σήμερα, μια και είναι η, η, η, η μέρα ε, για τις... Ε, σπάνιες ε, ε, ασθένειες. Ε, είναι σημαντικό έτσι ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση και γνώση αυτών των ανθρώπων που δεν ακούγεται είτε στο δημόσιο λόγο είτε στην έρευνα. Εδώ θεωρούμε ότι έχουμε πλέον μία σημαντική καμπή στο δικαίωμα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Ευρωπαίοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Ε, η κατάσταση όσων πάσχουν από σπάνιες ε, ασθένειες είναι περίπλοκη, μερικές φορές δε και δραματική. Ε, υπό τον γενικό ορισμό των σπανίων ασθενειών περιγράφονται ασθένειες οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικές εκφάνσεις και επομένως είναι θέμα σεβασμού προς τον ίδιο τον άρρωστο αλλά και τις οικογένειε των πασχόντων ε, το να ε, αντιμετωπιστεί ε, το ε, θέμα αυτό. Μην λησμονούμε ότι ο κανονισμός 141 έδωσε για τα ορφανά φάρμακα έδωσε την δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπείες σε ανθρώπους που δεν, είχαν καμία δεν είχαν διορθώνω καμία δυνατότητα θεραπείας. Αλλά θα πρέπει βεβαίως και στον τομέα της έρευνας, στον τομέα της... του συντονισμού των εθνικών πολιτικών να κάνουμε ε, οπωσδήποτε περισσότερα. Ε, υπάρχουν περιφέρειες όπως ας πούμε η Μεσημβρινή Ιταλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες που η στήριξη των πασχόντων από πλευράς του δημοσίου είναι σαφώς ελλειπής. Υπάρχουν κοινότητες ανθρώπων οι οποίες ζουν με μεγάλη δυσκολία, αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια για τη θεραπεία τους ε, αναγκάζονται να πηγαίνουν ε, σε κέντρα ή ακόμα και σε χώρες μακρινές ε, από τον τόπο διαμονής τους και αυτό οπωσδήποτε μειώνει και την εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λοιπόν τα προβλήματα που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ασθενείς. Σήμερα είναι η ημέρα λοιπόν των σπανίων ασθενειών και εάν αυτή η ημέρα έχει μία έννοια είναι ακριβώς για να μας θυμίσει ότι το δικαίωμα στην φαρμακευτική αρρωγή και το δικαίωμα στην θεραπεία πρέπει να είναι ίδιο δικαίωμα για όλους. Ευχαριστώ. Grazie, Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κύριο Πεδητσίνη. Συμμερίζομαι τα όσα υπόθηκαν ε, και βεβαίως πρωτοβουλίες όπως ε, η ημέρα ε, των ασπανίων ασθενειών είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί αποτελούν μια καλή ευκαιρία για πληροφόρηση των πολιτών. Έρχομαι στο προκείμενο. Ε, παρότι οι ασθενείς ε, που πάσχουν ε, από σπάνιες ασθένειες είναι λίγοι, το πρόβλημά τους είναι πολύ μεγάλο διότι ακριβώς επειδή είναι σπάνιες ασθένειες η έρευνα είναι μικρότερη, τα φάρμακα είναι λιγότερα, η πιο ακριβά, η πρόσβασή τους δύσκολη. Επίσης, ε, η φαρμακευτική ε, βιομηχανία δεν έχει ε, μεγάλο συμφέρον και ενδιαφέρον λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών να αναπτύξει φάρμακα. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις οι ασθένειες αυτές είναι ιδιαίτερος σοβαρές. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία παρουσιάζονται σε νεανικά νεανική, ε, βλέπε παιδική ηλικία ε, και επομένως ε, και σε όρους ψυχολογικούς και ψυχοκοινωνικούς είναι ιδιαίτερος επιβαρυντικές, επιβαρυντικές για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και για, τον, για την οικογένεια λόγω της γενούς δυσκολίας αλλά και των επιπλέον δυσκολιών ε, ε, αυτές ε, οι σπάνιες ασθένειες δεν θα πρέπει να γίνουν παραμελημένες ασθένειες. Αυτό είναι το σημαντικό και εάν η βιομηχανία δεν θέλει να αναλάβει το κόστος των, της έρευνας για φάρμακα για τέτοιες ασθένειες τότε θα πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς από τη δικιά μας πλευρά. Εμείς επανειλημμένα έχουμε προωθήσει την ιδέα Τη της δημιουργίας μιας φαρμακευτικής υπηρεσίας ε, που θα δίνει ε, χρήματα ε, που από μόνη της θα μπορεί να φτάσει σε καλά αποτελέσματα γιατί διαφορετικά έχουμε αυτήν την παράδοξη κατάσταση όπου η βιομηχανία θα βάλει χρήματα στην έρευνα μόνο εάν είναι σίγουρη ότι τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες σύντομες απαντήσεις στις παρατηρήσεις. Καταρχάς, διασύνδεση των ερευνητικών προγραμμάτων με τη δημόσια υγεία και τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Εδώ έχουμε κατευθυντήρες γραμμές για καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων δημόσιας υγείας, ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ε, κοινωνικής πρόνοιας και ασθενών από πασχόντων από σπάνιες ασθένειες. Είναι κάτι το οποίο καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν έξω από το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τι άλλες βελτιώσεις μπορεί να υπάρχουν στη διασύνδεση με, για τις ε, σπάνιες ασθένειες. Ο κ. Κατουτσίνη επίσης αναφέρθηκε σε προτεραιότητες για την έρευνα είπε ότι θα υπάρχει μια κοινή πρωτοβουλία για το 2019 προγραμματισμού που θα επιτρέψει τη συνεργασία σε προγράμματα ερευνητικά των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στόχευση συγκεκριμένα στις Ισπανίες νόσους. Ως προς την υλοποίηση της νομοθεσίας σχετικής με τα σπάνια φάρμακα και τα ορφανά φάρμακα και αυτά που ανέφερε η κυρία Γκροστέτ ότι πολλέ φορέ χρειάζεται οι ασθενεί να φύγουν από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε αλλού. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει. Θέλω να επισημάνω ότι η μέθοδος αξιολόγηση που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βελτιώσει την ε, προβολή και νέας τεχνολογίας ε, μεθόδων ε, θεραπευτικών, αλλά ταυτόχρονα και στο χώρο των φαρμάκων πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και έτσι έχουμε γενναίες κατευθυντήριες γραμμές ετοιμάσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκου πρόσβαση στα φάρμακα. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπό επεξεργασία μια έκθεση η οποία θα εξετάσει την πρόσβαση στα φάρμακα και τη δημολόγηση. Με πολύ ενδιαφέρον θα εξετάσουμε όταν βγει την έκθεση αυτή. Και βέβαια θα συνεχίσουμε και τις συζητήσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, για την πρόσβαση στα φάρμακα. Ε, έγινε αναφορά στο πρόγραμμα της Προεδρίας της Μάλτας και το ε, εργαστήριο μελέτης ε, το Μάρτιο για τις σπάνιες νόσους που θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για τους Υπουργούς να εξετάσουν ε, τα δεδομένα, τα προβλήματα και τη βελτίωση της πρόσβασης. Η κυρία Ντάλη αναφέρθηκε νομίζω στις τοποθετήσεις της σε μικρότερα κράτη-μέλη και εδώ πάλι τα δίκτυα αναφοράς 24 θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, θα αποτελέσουν μια πολύ χρήση, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο με προστιθέμενη αξία ιδιαίτερα για τα μικρότερα κράτη-μέλη και για τη συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας για την ε, ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ήθελε στο στάδιο αυτό να κάνει ή οδήποτε σχόλιο, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ακόμη η κοινοποίηση. Στο στάδιο αυτό ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε Πρόεδρο ολοκληρωνουμε εδω τη συζήτηση για σήμερα και την ημερήσια μας διάταξη. 9 Μαρτίου είναι η προσοχή μας, η συνεδρίαση και σας καλώ τώρα να κάνουμε μια ομαδική φωτογραφία. Έξω από την αίθουσα ο φωτόγραφος μας παρακάλεσε να βγούμε από την αίθουσα σε ένα κατάλληλο σημείο για να, πάρουμε, να κάνουμε αυτή τη φωτογραφία.